Συνήθω. Καλημέρα σε όλες και όλους σας. Εχθές είχαμε μια συνεδρίαση πάρα πολύ πυκνή και έντονη. Πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Και συνεχίζουμε σήμερα με αυτήν. Με μια συνεδρίαση εργασίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επίσης ε, διονγκωμένη, όπου έχει κυρίαρχο ρόλο ως δεύτερο σημείο η ψηφοφορία των γραμμών του προϋπολογισμού για το 2010 σε σχέση με τα θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων αρμοδιότητα αυτών, αυτής της Επιτροπής Ελευθεριών. Στις 9.30 θα γίνει αυτή η ψηφοφορία για να μπορέσουμε να έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό μελών παρόντων να μπορέσουν να συμμετάσχουν δηλαδή το δυνατόν περισσότερα μέλη. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι όμως η ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση που συντάσσει η Ευρωβουλευτήνα κυρία Ρενάτε Βέμπερ που έχει συντάξει για την πρόληψη δηλαδή και διευθέτηση επίλυση συγκρούσεων σε δικαιοδοσία ποινικών δικαστηρίων, ποινικέ διαδικασίες. Είναι η δεύτερη φορά που ζητείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει και να συντάξει μια γνωμοδότηση για αυτό το νομοθετικό θέμα ως πρωτοβουλία. Και ζητείτε τώρα από μας η έκφραση αυτής της γνωμοδότησης στην τελική αυτή φάση της εκπόνησης αυτής της απόφασης πλαισίου που βλέπουμε λοιπόν ότι στον τρίτο πυλώνα εντάσσεται όπου πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο και γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την έκθεση, την παρουσίαση της έκθεσης από την Ευρωβουλευτήνα κυρία Βέμπερ. Παρακαλώ κυρία Βέμπερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Αυτό το σχέδιο για την λήψη απόφασης είχε περιπετειώδη βίο μέχρι σήμερα. Είχε ξεκινήσει ως πρωτοβουλία διαφορετικών κρατών μελών υπό την ηγεσία της τσεχικής δημοκρατίας, της δημοκρατίας της Τσεχίας που ήταν, είχε τότε την Προεδρία ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου. Συντάχθηκε ένα σχέδιο έκθεσης, στη συνέχεια το Συμβούλιο εργάστηκε και ενέκρινε όμως ένα τελείως διαφορετικό κείμενο και ζητήθηκε να επαναδιαβουλευτεί το Κοινοβούλιο γι' αυτό και αυτό επεξηγεί γιατί το σχέδιο απόφασης πλαισίου βρίσκεται τώρα στο Κοινοβούλιο ως θέμα διότι με την νέα αυτή ε, διατύπωση πρέπει να υπάρξει νέα νομοδότηση. Θα είμαι πολύ πιο ήπια στην αξιολόγηση αυτή του, αυτής της απόφασης, σχεδίου απόφασης πλαισίου σε σχέση με την ε, αρμόδια επιτροπή για τα θέματα ποινικού δικαίου που είχε ζητηθεί γνωμοδότησή της από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαν ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί αυτή η πρόταση επειδή δεν προσφέρει τίποτα το καινούριο σε αυτό, για το θέμα αυτό. Ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε το κείμενο, το εξετάσουμε, πέρα από ένα μακρύ τίτλο, η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρούμε τίποτα για την πρόληψη συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικέ διαδικασίες που θα μπορούσε ίσως να διευθετηθεί με την ε, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και την αναγνώριση ε, αποφάσεων λόγω αυτής της ε, δικαιοδοσίας. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πει κανείς τι θα γίνεται σε σχέση με την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων δικαιοδοσίας. Για αυτούς τους λόγους η έκθεση που συνέταξα στρέφεται σε ένα αριθμό θεμάτων που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κείμενο θα μπορούσαν να το κάνουν πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό. Και εκφράζεται έτσι και η προσέγγιση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών κατά τη διάρκεια των ετών όσον αφορά την προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, όσον αφορά δικαιώματα κατηγορουμένων ή υπόπτων. Τώρα, έξι πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Έξι σημεία τα οποία θίγονται από την έκθεση που συνέταξα. Πρώτα, όπως είπα, το σχέδιο αυτό πρότασης δεν διαρθρώνει ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να επιλύει πραγματικά αυθεντικές συγκρούσεις δικαιοδοσίας ή συμφερόντων απλά δημιουργεί ένα είδος διαβούλευσης ή διεργασιών διαβούλευσης, αλλά όχι δεσμευτικά, ε, δεσμευτικών από πλευράς νομικής ή και προθεσμιών. Και ανέλαβα την πρωτοβουλία επίσης να επισημαίνω, να επισημάνω αυτά τα θέματα. Όμως πέρα από αυτά η μεγαλύτερη συνεισφορά παρέμβαση αυτής της πλευρά είναι η και προθεσμιων και ανελαβα την πρωτοβουλια επισης να να επισημανω αυτα τα θεματα ομως περα απο αυτα η μεγαλυτερη συνεισφορα παρεμβαση αυτης της εκθεσης ειναι η εμπλοκη της Eurojust για την πραγματική επίλυση τέτοιων προβλημάτων δικαιοδοσίας. Η Eurojust πιστεύω εγώ ότι είναι η καλύτερα τοποθετημένη, η καλύτερη υπηρεσία για να μπορέσει τέτοιου είδους θέματα να αναλάβει. Όχι μόνο σε εκείνους τους τομείς όπου έχει εξουσίες και αρμοδιότητες η Eurojust, δηλαδή σε διασυνοριακά σοβαρά εγκλήματα και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια σύγκρουση δικαιοδοσίας διότι απλά και μόνο με την αρχή του nec bis in idem θα πρέπει να δούμε ότι για την ε, ε, προσαγωγή στα δικαστήρια για δεύτερη φορά θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο ή πού θα μπορούσε να γίνει μια επανεξέταση, μια νέα δίκη. Ένα δεύτερο σημείο αφορά ένα μια ε, ειδοποίηση σε σχέση με τον ε, κατηγορούμενο. Πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής ε, ο, το, το, ως άτομο ο κατηγορούμενος. Όχι δηλαδή μόνο να ενημερωθεί για αυτή την πιθανή σύγκρουση δικαιοδοσίας, αλλά και για την συνολική κατάσταση και να έχει και δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, να προσφύγει δηλαδή κατά της λύσης που ε, θα υιοθετείται. Διότι πρόκειται ακριβώς για τα δικαιώματα της ή δικαιώματα του, της κατηγορουμένης ή κατηγορουμένου που διακυβεύονται εδώ. Επίσης τώρα σε σχέση με τον επίσημα κατηγορούμενο ως άτομο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα αυτού του ατόμου θα προστατεύονται. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το κείμενο όπως προτείνεται από τους συντάκτες αυτής της πρότασης είναι πολύ γενικόλογο και δεν ρυθμίζει αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε εδώ το θέμα των ε, προσωπικών δεδομένων που θα περιορίζουν αυστηρά στο όνομα επώνυμο διεύθυνση αυτού του ατόμου και όχι στην αποκάλυψη άλλων προσωπικών δεδομένων. Αρκετές τροπολογίες που θα βρείτε στην έκθεση αποσαφηνίζουν, αλλά διευκρινίζουν, αλλά και καθιστούν σαφές ότι μόνο δικαστικές αρχές είναι εκείνες που έχουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με θέματα συγκρούσεων δικαιοδοσίας. Καμιά άλλη αρχή, μόνο δικαστικές αρχές τι σημαίνει αυτό. Ένας ε, δικαστής, ε, ανακριτής δικαστής, ε, δημόσιος ε, εισαγγελέας λοιπά, Κατήγορος εισαγγελέας λοιπά. Με αυτή την σύντομη παρουσίαση θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό το σχέδιο πρότασης δεν ρυθμίζει τις πτυχές των αρνητικών συγκρούσεων δικαιοδοσίας. Και έτσι θα έλεγα ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να διευθετήσει αυτό το θέμα. Κάτι να γίνει σχετικά χθε. Για, σας, για εκείνους από εσά που συμμετείχατε στην αίθουσα, ζήτησα από την Σουηδέζα Υπουργό Δικαιοσύνης όσον αφορά κάποιες ασύμβατότητες μεταξύ αυτού του κειμένου και άλλου σχεδίου όσον αφορά την ε, μεταβίβαση ε, των ε, διεργασιών δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις πλαίσιο αλλά θα πρέπει να είναι συμβατές η μία με την άλλη. Η μία όσον αφορά τις διεργασίες και την μεταβίβασή τους όσον αφορά τα ποινικά θέματα που είναι έχει πολύ καλύτερα συνταχθεί και υποβάλει προτάσεις για λύσεις και όταν πρόκειται για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι πολύ καλύτερη στην σύνταξή της. Τούτη εδώ θα έπρεπε να τροποποιηθεί ή δυνατόν αν γίνεται από το Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Μου φαίνεται ότι το Συμβούλιο για κάποιους λόγους βιάζεται να εγκρίνει και να προχωρήσει. Είναι όμως από την άλλη πλευρά σημαντικό η Ευρωβουλή να υιοθετήσει την γνωμοδότηση αυτή στις γραμμές που εγώ σας εξέθεσα, ώστε τουλάχιστον να αποσταλεί ένα μήνυμα στο Συμβούλιο για το ποιο είδους λύση εμείς ε, έχουμε, ποια είδους λύση έχουμε υπόψη όταν κάνουμε λόγο για την ε, επίλυση θεμάτων συγκρούσεων δικαιοδοσίας. Και έτσι ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια ανταπόκριση από τα άλλα όργανα. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σχόλια κάποιος που θέλει να παρέμβει. Εσείς παρακαλώ. Ναι, σημειώνουμε. Εντάξει. Η κυρία Λάτφορντ, παρακαλώ λοιπόν. Sorry, to jump ahead of... Δεν ήθελα <clears throat> να πάρω το λόγο πριν από τους σκιώδεις εισηγητές, δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βέμπα για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει. Τα σχόλια της συγκεκριμένη Επιτροπής σε επίπεδο ουσίας νομίζω είναι ακόμα πιο έντονα από αυτά τα οποία μας είπε. Για το τελευταίο σημείο το οποίο έθεσε η κυρία Βέμπερ, αν δεν υπάρχει συνεκτικότητα ανάμεσα στις ε, διάφορες διαδικασίες οι οποίες ε, αφορούν την μεταφορά των δικαστικών δεδομένων είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό των δικογραφιών από τη μία χώρα στην άλλη. Τι κάνει το Συμβούλιο. Περιμένουμε επιτέλους να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας έτσι ώστε τουλάχιστον στα ποινικά να μπορούμε να ακολουθήσουμε τις κανονικές νομοθετικές διαδικασίες με μεγαλύτερη διαφάνεια, διαφάνεια η οποία θα βοηθήσει τις σωστές αξιολογήσεις και θα λύσει ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Και τα ακούσαμε χτες από τον πρόεδρο του Eurojust. Μας, είπε, μας έδωσε μια εικόνα της κατάστασης η οποία είναι πράγματι εκτρή. Διερωτώ λοιπόν ποια είναι η ποιότητα των εργασιών του Συμβουλίου εφόσον δεν στέκονται ικανοί να προσδώσουν μια κάποια συνεκτικότητα στις εργασίες αυτές. Και για τα άλλα σημεία τα οποία θέτει συμφωνώ μαζί της και τα υποστηρίζω. Κάποιες από τις προβλέψεις της νομοθετικής πρότασης είναι ιδιαιτέρως γελία εξασθενημένες. Λέγεται σε ένα σημείο σαν παράδειγμα ότι η απάντηση σε μία αναφορά θα πρέπει να δίδεται χωρίς ε, ε, υπερβολική καθυστέρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τι θα πει αυτό. Μα είπαν εχθέ στα πλαίσια τη παρουσίαση τη ετήσια έκθεση του Eurojust ότι μία απάντηση σε μία τέτοια αναφορά μπορεί να απαιτήσει δύο ολόκληρα έτη. Δεν υπάρχει ουσιαστική προθεσμία, δεν υπάρχει ουσιαστικός χρονικός περιορισμός. Θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, ε, ορισμού μιας χρονικής προθεσμίας, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα μια τέτοια απάντηση. Σχετικά τώρα με την τροπολογία 14. Αντί για αυτήν την ιδιαίτερα, θα έλεγα, χαλαρή διατύπωση, η οποία λέει ότι οι υπηρεσίες των κρατών μελών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα τα οποία θεωρούν ότι είναι σχετικά με την υπόθεση. Δεν λέει τίποτα αυτή η φράση. ενώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λάβουν ε, οι εθνικές αρχές υπεύθυνα υπόψη. Και η κυρία Βέμπερ έχει φυσικά πολύ δίκιο όταν καθιστά την διαβούλευση και την εμπλοκή του Eurojust ουσιαστικά υποχρεωτική, κάθαρη μάλλον, πολύ συγκεκριμένη. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η ισχύουσα πρόταση λέει ότι θα πρέπει διαβουλεύσεις οι οποίες δεν θα αποκλείουν την δυνατότητα επαφής και εμπλοκής του Eurojust. Τι, θέλει να πει αυτή η φράση. Πραγματικά είναι εντελώς χαλαρή, εντελώς παθητική φράση, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί το έχουμε το Eurojust αν δεν το χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τι είδους διασυνοριακή συνεργασία θέλουμε. Δεν ζητάμε να υπάρξουν αλλαγές στα εθνικά νομικά συστήματα. Θέλουμε απλά να καταστήσουμε μεταξύ τους τα εθνικά νομικά συστήματα ικανά να επικοινωνήσουν, να αλληλοεπιδράσουν το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, όλο και περισσότερες προτάσεις γίνονται για συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων, στοιχείων, αλλά σε επίπεδο εντελώς βασικό. Η συνεργασία ανάμεσα στα νομικά συστήματα, στις εθνικές δικαιοδοσίες δεν υπάρχει ή αν υπάρχει δεν εφαρμόζεται, δεν μεταφέρονται οι διατάξεις οι οποίες ισχύουν με σωστό τρόπο. Το Συμβούλιο λοιπόν είναι υπόλογο για αυτή την κατάσταση και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το λάβουν υπόψη τους γιατί έχουν αποτύχει στο Συμβούλιο να δώσουν λύσεις μέχρι τώρα. Και η Ρενάτε έχει απόλυτα δίκιο όταν υπογραμμίζει τις λεγόμενες διαδικαστικές εγγυήσει. Δεν θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις να γίνονται εν αγνία αυτών οι οποίοι είναι οι πρώτοι θα έλεγαν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση, να είναι ενήμεροι, να κάνουν αναφορές, να παρεμβαίνουν στις διαδικασίες, να ζητούν αλλαγή δικαιοδοσίας ή τουλάχιστον να προτείνουν την δικαιοδοσία, την νομική, η οποία θεωρείται η καλύτερη και η καταλληλότερη για κάθε περίπτωση. Ελπίζω να υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη Σουηδική Προεδρία γύρω από όλα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Λούτφορντ. Υπάρχουν και άλλα μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Θυμίζω ότι στις 9.30 έχουμε την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω για μια ακόμη φορά να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά παρακαλώ. Μακοβέη. ορίστηκα σκιώδης εισηγήτρια από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάρα πολύ σύντομα τα μέτρα τα οποία προτείνονται στα πλαίσια αυτής της πρότασης απόφασης έχουν σαν στόχο την αποφυγή του να διώκεται κάποιο σε δύο διαφορετικές χώρες για τα ίδια γεγονότα. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις των μίντεμ και να αποφύγουμε επίσης για δικαιολόγητες καθυστερήσεις οι οποίες προέρχονται από τη χρήση μέσων και στοιχείων από δύο διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες. Δεν θα πρέπει κάποιος φυσικά να δικάζεται για το ίδιο γεγονός δις. Υπάρχει όμως μια διαφωνία γύρω από το ποιος θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, την δικαστική και την προανακριτική διαδικασία. Αυτές οι διαφωνίες δυστυχώς προκαλούν καθυστερήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια σημεία έτσι ώστε να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις αυτές και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ακριβέστερες προτάσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε παρανεώσεις στο μέλλον και ερμηνείες οι οποίες θα δημιουργούν συγχύσεις και δεν θα διευκολύνουν την απονομή της δικαιοσύνης και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων πολιτών. Καλωσορίζω την ιδέα να υπάρχουν προθεσμίες χρονικές για τις διαδικασίες αυτές και να υποχρεώσουμε ουσιαστικά τις αρχές να απαντούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Θα καταθέσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την αποτελεσματικότητα της απονομής δικαιοσύνης. Ένα παράδειγμα. Οι λεγόμενες παράλληλες δικαιοδοσίες οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των διαδικασιών των δικαστικών, αλλά για τα προδικαστικά, ιδιαίτερα στην αρκτική φάση μιας ανάκρισης, μιας προανάκρισης δηλαδή, και στην περίπτωση που οι αστυνομικές αρχές είναι υπεύθυνες για τις προανακριτικές διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ενημέρωση έτσι ώστε να αποφεύγονται ε, επικαλύψεις και καθυστερήσεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Επαναλαμβάνω ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες στα πλαίσια των προθεσμιών τις οποίες μας προτείνατε. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Η προθεσμία, σας θυμίζω, για την κατάθεση των τροπολογιών για την έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι η 9η Σεπτεμβρίου. Θα το έλεγα στο τέλος της συζήτησης, αλλά έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Άλμπρεχτ. Θα είμαι σύντομος. Η έκθεση βαδίζει την σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται εννέα συστήματα αντί να υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές νομικής προστασίας. Γιατί είναι σωστό να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές για αυτούς που ε, ενδεχομένω υφίσταται δίωξη. Και για μια αμοιβαία αναγνώριση που εάν λείπει μπορεί να είναι αντιδημοκρατική. Χρειαζόμαστε πάντως ελάχιστες προδιαγραφές, χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφές νομικής προστασίας στις οποίες να μπορούν να αναφέρονται οι πολίτες και αυτό θα είναι εγγυημένο μόνο εάν υπάρχει ευθεία πρόσβαση. Για παράδειγμα, να μην υπάρχουν γλωσσικοί φραγμοί, ώστε τα δικαιώματα των πολιτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων να μπορούν οι πολίτες να τα αξιώνουν ευθέως. Και γι' αυτό μας ικανοποιεί εν τέλει η έκθεση. Δεν υπάρχουν πλέον σχόλια. Καλό θα ήταν να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ λοιπόν η εκπρόσωπος της Σουηδικής Προεδρίας, νομίζω ότι πρέπει να είναι εδώ, ή ο εκπρόσωπος, έχετε το λόγο, όχι. Άκουσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον την συζήτησή σας και θα επιδιώξουμε να λάβουμε υπόψη μας την άποψη του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της τελικής απόφασης για τις αντιτιθέμενες ε, δικαιοδοσίες και τις διαφωνίες που μπορεί να προκύπτουν. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό και στα πλαίσια της παρουσίασης την οποία έκανε χθε η Υπουργός κυρία Άσκ χτες το πρωί. Αναφέρθηκε η κυρία Άσκα και στις διασυνδέσεις που έχει αυτή η πρόταση για απόφαση και με άλλες προτάσεις οι οποίες είναι υποσυζήτηση στο Συμβούλιο σε αυτή τη φάση. Φυσικά δεν έχουν όλες τον ίδιο στόχο, συμπληρώνουν η μία την άλλη και όπως είπε και η Βαρόνι Λόντφορντ, είναι ένα θέμα το οποίο θα προωθήσουμε αυτό σε σχέση πάντα και σε συνεργασία με αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων. <clears throat> Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προτάσή της. Θα την εξετάσουμε λεπτομερέστερα σχετικά με την πρόταση για την απόφαση πλαίσιο. Υποστηρίζουμε τις γενικές γραμμές της πρότασης αυτής. Θα πρέπει να θεωρηθεί όμως η πρόταση αυτή σαν ένα πρώτο βήμα για την πρόληψη των διαφωνιών ανάμεσα σε διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει σε υστερότερη φάση μια πολύ λεπτομερέστερη πρόταση για την αποφυγή αυτών των επικαλύψεων. Yes, again, Mrs. Weber for concluding remarks. Uh, Κλείνει τη συζήτηση η κυρία Βέμπερ. Θα πρέπει να ορίσουμε την προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών και θα πρέπει να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους Κιώδης για να ορίσουμε τελικά την άποψη της ε, Επιτροπής μας. <clears throat> για μια ακόμη φορά λοιπόν θυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση ΒΕΜΠΑ είναι η 9η Σεπτεμβρίου. Έχετε μία εβδομάδα ακόμα λοιπόν και τις πρώτες, έχετε μάλλον τις υπόλοιπες μέρες αυτής της εβδομάδας και τις πρώτες της επομένης. Καλώς, σας ευχαριστώ. Yeah. <laughs> As announced, there comes the time to proceed on the vote of the budgetary lines. I think we have worked. Θα συνεχίσουμε τώρα με την ψηφοφορία του προϋπολογισμού. That we can proceed now to vote on every amendment, but I understand. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουμε κάθε μία από τις προϋπολογίες. Αν καταλαβαίνω καλά υπάρχει όμως ένας διαδικαστικός κανόνας τον κανονισμό μας ο οποίος ε, μας διευκολύνει πολύ. Επειδή εγώ ήμουν εισηγητής, είχα διοριστεί σαν εισηγητής για την πρόταση που νομοδότησε για τις γραμμές του προϋπολογισμού, θα αντικατασταθώ στη συγκεκριμένη αυτή φάση και θα προεδρεύσει τη ψηφοφορία σε ένας άλλος συνάδελφος. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Ιντεβελτ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 μου, θυμίσουν, μου θυμίζουν ότι θα πρέπει να παρακαλέσω όλες και όλους να ενθέσουν τις ηλεκτρονικές κάρτες τους ε, στην σχισμήν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην ξεχάσετε να βάλετε την κάρτα σας λοιπόν. Η ε, κυρία Λάτφορντ. Δυστυχώς ξέχασα. Έχω την παλιά μου μαζί. Μήπως μπορείτε να σημειώσετε την, ε, τον τρόπο που θα ψηφίζω. Είναι το ίδιο. Διέθετε μέρα παρακαλώ. Ναι πρόεδρε. Έχω το ίδιο πρόβλημα όπως η κυρία Λάτφορντ. Δηλαδή, όπως και η δική μου πολιτική ομάδα παρακαλώ, να ληφθεί υπόψη ότι ψήφισα. κύριος Μπουσούτιλ. Uh, Φαίνεται ότι ορισμένα από τα μέλη δεν έχουν τις κάρτες τους. Σας παρακαλώ να σημειώσετε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν. ο Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχει διαδικαστική ένσταση, τότε είναι εντάξει. This I so I should, I should, I should go somewhere else? No, you can stay here. Si, uh, Irina, you come here. Irina, you come here. Will do I vote?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 Let's start uh, the voting. Good morning, everybody. Um, Η Προεδρεύουσα. Βλέπω ότι έχουμε πολλές σελίδες ε, για ψηφοφορίες. Εάν συμφωνείτε, διακόπτει μια κυρία. Γιατί? Δεν λειτουργεί. Καλώς. Εάν συμφωνείτε, μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες που επαναφέρουν το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2010 με εξαίρεση των τροπολογιών εκείνων, των κονδυλίων εκείνων, όπου έχουν κατατεθεί πλήρωνε τροπολογίες. Εάν συμφωνείτε, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη σελίδα 5. Παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι αν συμφωνείτε να ψηφιστούν όλες μαζί οι τροπολογίες που προανέφερα. Είναι σαφή η πλειοψηφία. Τώρα, η ερώτηση είναι ψήφι, ποιοι είναι υπέρ, ψήφοι υπέρ λοιπόν, της, των κονδυλίων όπου ε, επανέρχεται το ε, προσχέδιο του προϋπολογισμού. Δηλαδή μέχρι την σελίδα 5. Ψήφι υπέρ αυτών των κονδυλίων. Κατά. Και ποιος απέχει, Μία αποχή λοιπόν. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην σελίδα 5 του εγγράφου. Στην γραμμή 18-02-03-01. Τροπολογία ΛΥΜΠΕ 56-56. Θα αναφέρομαι τώρα στον αριθμό των τροπολογιών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Άρα 56-56 Στη σελίδα 5. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 56-52. Υπέρ. Κατά. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα όποιο έχει κάρτα να ψηφίσει και όσοι δεν έχουν θα ψηφίσουν σηκώνοντα το χέρι. Θα με βοηθήσετε κύριε Γραμματέα. Ναι, λοιπόν, μιλούμε για την 56-52. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μείνε με ηλεκτρονικές κάρτες, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε ποιος είναι υπέρ.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 Ας κλείσουμε την ψηφοφορία και θα δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Πρόκειται για τεχνική ψηφοφορία για να δούμε πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί καλά το σύστημα. Βλέπετε τίποτε. Ωραία. Επανερχόμαστε. Ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Για παράδειγμα, και το δικό μου μηχάνημα δεν λειτουργεί, αλλά και άλλα από κάτω από ό,τι βλέπω. Θα μετρήσουμε λοιπόν. Δεν διευκολύνει το έργο μας αυτό. Υπάρχουν πολλά μηχανήματα τα οποία δεν λειτουργούν. Καλώς. Άρα, αρχίζουμε ξανά. Τροπολογία 56-52 υπέρ. 25 υπέρ. Κατά. Είκοσι κατά. Αποχές. Καλά. Δεν έχει. Ωραία. Ακολουθεί 56-43 υπέρ. Για την προηγούμενη 56-52 έγινε ε, δεκτή με 25 υπέρ 22 κατά. Τώρα, 56-43 υπέρ. Καλώς. Απορρίπτεται. Α, όχι. Κατά, λέει η πρόεδρος. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. 56-48 υπέρ. Εκπίπτει εφόσον γίνει δεκτή 43. Κατά, παρακαλώ, τώρα συντούτην εδώ. Εγκρίνεται. 56-64. Μόνο τα σχόλια. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56-58. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 56-64. Είκοσι υπέρ, 23 κατά. 56-58. Υπέρ. Υπέρ είπαμε πρώτα. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 56-44. Εδώ έχει ζητηθεί μια ψηφοφορία κατά τμήματα για τους αριθμούς. Άρα πρώτα θα ψηφίσουμε τους αριθμούς. Ε, αν συμφωνείτε δηλαδή, να αυξηθούν κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, αντί 5. Το CA και PA. Ψηφίζουμε, ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται μάλιστα σαφώς. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα τα 5 εκατομμύρια. Ο αριθμός των 5 εκατομμύριων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα τα σχόλια. Υπέρ. Κατά. Ωραία, εγκρίνονται και αυτά. 56-12. Α, αυτό εκπίπτει. 56-66. Μόνο τα σχόλια. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μπουσουτίλ. Μπορείτε, παρακαλώ επιμένω, να ανακοινώσετε το αποτέλεσμα, ώστε όλοι να είμαστε καθυσυχασμένοι, να γνωρίζουμε τους ακριβείς αριθμούς. 20 υπέρ 22 κατάλληλοι πρώτος. πρόεδρος. Υπέρ. κατά 25 υπέρ 26 κατά. Πάμε πολύ σιγά έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με την ε, τεχνολογική πλευρά του θέματος. Γιατί υπάρχουν τα μηχανήματα. Yes, εκφράζω την ανησυχία μου, διότι από το ένα λεπτό στο άλλο, μια ψηφοφορία που έδινε 20-22, τώρα δίνει 25-26. Ας προσπαθήσουμε ξανά να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό μηχάνημα και ας καταμετρούμε μόνο τις ε, ψήφους εκείνων των προσώπων που δεν λειτουργεί στο μηχάνημά τους. Ναι, και Κόπ. Η εξήγηση κύριε Μπούσουτιλ είναι ότι δεν ε, συμπεριλάβατε τις αποχές στις τελευταίες φοφορίες. Και με όλο τον απαραίτητο σεβασμό σας προτείνω να το κάνετε. Γι' αυτό ε, εμφανίζεται αυτή η διαφορά. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση. Αλλά παρακαλώ και εγώ να συνεχίσουμε. Ιακολίνο. 42 πήραν μέρος στην ψηφοφορία σε σχέση με τους 51 οι οποίοι ψήφισαν την επόμενη φορά. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά μπήκαν 11 άτομα βιαστικά από τη μία στιγμή στην άλλη στην αίθουσα. Και αναφέρομαι στην ψηφοφορία των τροπολογιών 566 και 567. Παρακαλώ θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς ε, διεξάγεται η ψηφοφορία και τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα. We should try to check it electronically. Θα προσπαθήσουμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά ηλεκτρονικά. Έχουμε τις δύο αυτές τροπολογίες οι οποίες πράγματι ήταν αμφίροπη η ψηφοφορία και στις δύο. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε όμως στις ψηφοφορίες αυτές. 56-66 και μετά 56-67 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πρώτα την 56-66.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 47 κάρτες λέει η πρόεδρος, από τις οποίες ε, λειτουργούν οι 42. Από αυτές τις 42, 16 ψήφισαν υπέρ, 24 ψήφισαν κατά. Τώρα, ε, όσοι δεν δουλεύει η μηχανή τους να σηκώσουν τα χέρια τους παρακαλώ. Να ψηφίσουν διανατάσεως. Αν το φωτάκι, η λάμπα στο μηχάνημά σας είναι πράσινη, σημαίνει ότι δουλεύει. Αν είναι κόκκινη, σημαίνει ότι δεν δουλεύει και θα ψηφίσετε δια ανατάσσεως χειρών. Λοιπόν, 19 υπέρ συνολικά και τώρα πόσοι είναι κατά και 26 είναι κατά, 16, 19 συγγνώμη είναι υπέρ και 26 είναι κατά και δύο αποχές. Συνεπώς η 56-66 απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 5667. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 56-67. Τέλος. Και τώρα θα ψηφίσουν σε εισαγωγικά οι χειρονάκτες. Είκοσι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. 28 κατά. Δεν έχουμε αποχές στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνεπώς απορρίπτεται η 56-67. Φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική υπαρίθμου 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απέχουν. Δεκτό. 56-68. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5668. Τέλος ψηφοφορίας. Ποιοι είναι παρακαλώ υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ των οποίων θυμίζω δεν δουλεύει το μηχάνημα. «22 είναι υπέρ, συνολικά. Ποιοι είναι κατά. «26 κατά. Ποιοι απέχουν δεν υπάρχουν αποχές, απορρίπτεται. Η 56-68. Φτάνουμε τώρα στην 56-14. Και είναι υπέρ. 56-14. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56-14 παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Ποιοι είναι υπέρ. Υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία. Τώρα 56-69. Ποιοι είναι υπέρ. Και εδώ χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 56-69. Θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά από εδώ και πέρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πέντε συνάδελφοι των οποίων δεν δουλεύουν οι κάρτες. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 5669. Δεκαεπτά υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. Τώρα φτάνουμε στην προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Η ηλεκτρονική ψήφος. Τέλος της ψηφοφορίας για την προφορική τροπολογία. 25, κατά 25 υπέρ 17 κατά γίνεται δεκτή η προφορική. Τώρα η 56-77 αποσύρεται. Η 56 καταπίπτει. Η 56.78 ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56.78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 Sí. Queridos colegas, por favor. Como saben, estamos muy constreñidos en la gestión del tiempo porque... Για την ε, διαχείριση του χρόνου αμέσω, μετά από αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη θα έχουμε μια συνεδρίαση διμερή με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε τη διαδικασία SWIFT. Και γι' αυτό ζητώ κατανόηση λοιπόν από πλευρά σας, διότι θα ακούσουμε τώρα σε σχέση με την έκθεση του συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, υλοποιώντας τους στόχους της αντιτρομοκρατικής ε, πολιτικής, στο, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ζητώ κατανόηση λοιπόν λέω, διότι στη διαχείριση του χρόνου θα ακούσουμε βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή του, αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε γύρω συζήτηση αμέσως μετά την εισήγησή του. Έτσι τα, μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών καλούνται να διατυπώσουν γραπτώς ερωτήσεις και παρατηρήσεις που θα έχουν στην εισήγηση, στην έκθεση που θα ε, έχουμε για να μπορέσουμε λοιπόν ιστερότερα, μεταγενέστερα να προβούμε στην εξέταση του ε, θέματος SWIFT που συμπεριλαμβάνει το σύνολο αρχών και φορέων εσωτερικών και εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν για αυτή την ακρόαση, για αυτό το θέμα. Και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση <clears throat> έχουμε τον συντονιστή ενώπιόν μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιλντε Κέρκοφ, που προσέρχεται για πρώτη φορά σε αυτή την πολιτική κοινοβουλευτική επιτροπή πολιτικών ελευθεριών μετά την ε, συγκρότηση του νέου κοινοβουλίου. Τον καλωσορίζουμε, του ευχόμαστε την καλύτερη επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων του. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Πάντα θέλω να έχω στενές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την δική σας Επιτροπή. Για προφανείς λόγους, γιατί η πρόληψη και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εμπλέκει και τα κοινοβούλια των χωρών μελών και φυσικά το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ιδιαίτερα με δύο από τους ε, προηγούμενους προέδρους αυτής της Επιτροπής και είμαι ανυπόμονος εκ νέου να ξεκινήσουμε ένα ποιοτικό διάλογο, ένα ισότιμο διάλογο και με σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος για να επιτρέψω να υπάρξει μια κάποια συζήτηση η οποία θα μου είναι ιδιαίτερο χρήσιμη και είμαι στη διάθεσή σας και για γραπτές ερωτήσεις. Να πω ότι παράλληλα με την ΕΤΑ και αναφέρομαι στα, στα απόπειρε της καλοκαιρινέ του Μπούργο, την δολοφονία δύο χωροφυλάκων στην Πάλμα Μαγιόρκα στο τέλο Ιουλίου και να σημειώσω εδώ και μια πολύ καλή γαλλο-ισπανική συνεργασία που οδήγησε στην ανακάλυψη μιας κρύπτη όπλων. Παράλληλα με όλα αυτά, ο Ισλαμικός ακραίο ε, η ακραία τρομοκρατία απειλεί πάντα απειλεί την ασφάλεια των κρατών μελών, των πολιτών μας, αλλά και των α, συμπολιτών μας όταν μετακινούνται στο εξωτερικό. Βέβαια από την εποχή του Λονδίνου δεν υπάρχουν άλλες τέτοιες απόπειρες. οι, αντι... οι υπηρεσίες ασφαλείας γενικά έχουν καταφέρει να αποτρέψουν πολλές επιθέσεις και απόπειρες, αλλά παρόλα αυτά ε, θα ήταν λάθος να πιστέψει κανείς ότι το επίπεδο απειλής έχει πράγματι χαμηλώσει. Η αλήθεια είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χαμήλωσε το επίπεδο, θα έλεγα, συναγερμού, αν και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, σύστημα ταξινόμησης αριθμητικό ή με χρώματα. Παρ' αυτά, Υπάρχει το θέμα της δεξαμενής, θα έλεγα, έβρεσης προσώπων για την τρομοκρατία που παραμένει. Καταρχάς, να σταθώ ε, στην τρομοκρατία σε σχέση με φαινόμενα εξέγερσης. Το δεύτερο είναι κάποιες χώρες ε, οι οποίες καθίστανται όλο και πλέον έφραστες. Το Πακιστάν, σαν παράδειγμα, η Εμένη, οι χώρες του Σαέλ, και το είπε ο Γάλλος πρόεδρος αυτό στην ομιλία που έκανε προς τους διπλωμάτες του και όλα αυτά επιτείνονται από την οικονομική χρήση και μετατρέπονται κάποιες τέτοιες χώρες σε καταφύγιο της Αλκάιντα στα πλαίσια ενός φαινομένου περιφερικοποίησης της Αλκάιντα. Υπάρχει Αλκάιντα στο Μαγκρέμπ, στο Σαέλ, στη Μεσοποταμία, στην Αραβική Χερσόνησο. Ένα δεύτερο φαινόμενο είναι ο αριθμός των Ευρωπαίων που πηγαίνουν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Οι αριθμοί από ό,τι φαίνεται είναι ψηλοί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρόσφατη περίπτωση και να καταλάβετε ε, σε τι αναφέρομαι. Η Ιταλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2008 δύο Γάλλων δύο Γάλλων οι οποίοι ε, διευκόλυναν κάποιους παράνομους μετανάστες. Ε, φάνηκε από την έρευνα ότι ήταν σημαντική υπεύθυνη στελέχη της Αλκάιντα, προέβλεπαν απόπειρε στη Γαλλία και στην Αγγλία και ήταν μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου και λειτουργούσαν κάνοντας προπαγάνδα μέσω του διαδικτύου. Ο ένας Συριακής εκπαίδευσης ήταν υπεύθυνο για το Βελγικό Ισλαμικό Κέντρο και μέσω του κηρύγματός του προωθούσε την Ισλαμική προπαγάνδα. Ο άλλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνο πληροφορικής, ήταν υπεύθυνο επίσης μιας ιστοσελίδας υπέρ της τζιχάτ και της βίας. Και στήριζαν ένα δίκτυο τζιχαντικό ε, το οποίο τροφοδοτείται από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Παρ' όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία αυτού του φακέλου, δηλαδή σύλληψη στην ε, Γαλλία ε, Ιταλών ή μάλλον στην Ιταλία Γάλλων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ε, το ίντερνετ, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για παράνομες μεταναστεύσεις τελεχών από και προς το Πακιστάν. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν θα έλεγα το πόσο στοχευμένη σωστά είναι η στρατηγική την οποία υθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2007. Το θέμα δεν είναι να αποκαλύψουμε μόνο ε, τα δίκτυα αυτά, αλλά να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε σωστά και με συνεχή τρόπο τους τέσσερις άξονες της στρατηγικής αυτής, δηλαδή πρόληψη, ανταπόκριση, παρακολούθηση και κατευνασμός. Αυτά όλα περιλαμβάνονται και στο έγγραφο συζήτηση το οποίο έχει διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποια επιμέρους στοιχεία. Ο πρώτος άξονας των εργασιών μας και νομίζω ότι είσαστε κι εσείς ιδιαίτερα δραστήριση σε σχέση με αυτό είναι το θέμα της συλλογή και κυκλοφορίας της πληροφόρησης. Εδώ και δύο χρόνια προσεκάλεσα το Συμβούλιο να ξεκινήσει τον ορισμό μιας στρατηγικής συλλογής πληροφοριών. Σημερίζομαι πλήρως την τις θέσεις τις οποίες είχατε και πριν από τις ευρωεκλογέ και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τώρα την αίσθηση που έχετε ότι το Συμβούλιο προχωρά με εμπειρικό τρόπο, πολλαπλασιάζοντας τα σχέδια και τα προγράμματα, χωρίς να έχει μια συνολική όμως άποψη για την στρατηγική και για την απόσταση την οποία θέλουμε να διανύσουμε στα πλαίσια των μεθόδων συλλογής πληροφοριών. Και στα πλαίσια της εκθέσεως την οποία έχω προσαρτήσει κάνω ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές από το πρόγραμμα της Στοκόλμης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε κάποιους ορισμούς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τις εργασίες μας συνεκτικότερες. Δεν θα ήθελα να περάσω σε λεπτομέρειες. Η Ευρωπόλ και η Ευρωτζάστα έχουν εμβαθύνει την συνεργασία την οποία είχαν μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει πρόοδος που πρέπει να γίνει. Το πρόγραμμα Check the Web, έλεγχος του ιστού έχει προχωρήσει και αυτό αρκετά. Το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Είναι ένα θέμα το οποίο για πολλούς λόγους είναι δύσκολο να προωθήσει κανείς. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε κάποιες μεθόδους για να προσδώσουμε μια κάποια δυναμική στο πρόγραμμα αυτό, ε, δεχόμενοι κάποιες ε, χώρες πιλότους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και θα μπορούσαν να ασχοληθούν ειδικά με ένα από τα θέματα της στρατηγικής πρόληψης την οποία έχουμε και να συμμεριστούν τα συμπεράσματά τους με τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν 6-7 χώρες ε, μέλη σήμερα που ασχολούνται με ένα θέμα. Το Βέλγιο και η Σουηδία σαν παράδειγμα ασχολούνται με το θέμα τους εκ, του σύνεγγης αστυνόμευσης. Η Ολλανδία ασχολείται με το θέμα του ρόλου των τοπικών αρχών και συνεργάζομαι και με την Επιτροπή των Περιφερειών για το θέμα αυτό οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ε, να δώσουν κάποιες πρώτες απαντήσεις. Με τη Δανία επίσης συζητάμε το θέμα αυτό, με την Ισπανία είναι ευαίσθητο θέμα, είναι η κατάρτιση των θρησκευτικών ηγετών, των ημάμιδων. Με την Γερμανία το θέμα του διαδικτύου και με άλλες χώρες ε, τα θέματα επικοινωνίας μας και επαφής μας με τον Ισλαμικό κόσμο. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο δεν θα αναπτύξω είναι η εξωτερική πλευρά. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνω εδώ και αρκετού μήνε. Χαίρομαι για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενό συγκεκριμένου προγράμματο στα πλαίσια του μέσου σταθερότητα που βοηθά τι τρίτε χώρε, χώρε οι οποίε είναι θύματα φαινομένων τρομοκρατικών, να ενισχύσουν τι εσωτερικέ του διατάξει και τα εσωτερικά του μέτρα. Αυτό είναι ο πρώτο άξονα τον οποίο ακολουθήσαμε, ο δεύτερο άξονα. Και πηγαίνει αρκετά καλά εδώ η υπόθεση. Να δούμε με ποιο τρόπο Ξέρω ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Με ποιο τρόπο να βρούμε περισσότερα χρήματα στα πλαίσια της συνεργασίας για την ανάπτυξη και να καταλήξουμε σε προληπτικά μέτρα στις χώρες οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από το τρομοκρατικό φαινόμενο και αυτό κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χώρες του ΣΑΕΛ. Είδαμε ποιε ήταν οι ανησυχητικέ εξελίξεις το καλοκαίρι στη Μαυριτανία. Στο Μαλί έχει φαινόμενα αντίστοιχα να αντιμετωπίσει και γι' αυτό αυτά τα δύο τόξα κρίσης στην Δυτική Αφρική από τη μία συνδυασμός λαθρεμπορίου ναρκωτικών και, και οργανωμένου εγκλήματος σε χώρες όπως η Γουινέα Μπισάου και η κρίση στο ΣΑΕΛ δεν θα θέλαμε αυτά τα δύο τόξα κρίσης να έλθουν σε επαφή και να συναντηθούν και να συντονιστούν. Εργαστήκαμε επίσης για άλλα θέματα όπως το Πακιστάν τις τελευταίους μήνες για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το Πακιστάν να περάσει από μια στρατιωτική αντιμετώπιση του τρομοκρατικού φαινομένου που να βασίζεται σε μια πιο κλασική αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω των αστυνομικών αρχών και των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία στην έκθεσή μου σχετικά με τα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σχετικά με την έρευνα για τα θέματα ασφαλείας, για την ανάγκη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει περαιτέρω μέτρα στα πλαίσια της προστασίας του κυβερνοχώρου, επίσης και για τους κινδύνους βακτηριολογικού, χημικού και πυρηνικού ε, τρομοκρατικού φαινομένου. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία με απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό. Πρώτα, μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε στο Συμβούλιο για την ευρωπαϊκή ανταπόκριση σε κάποιες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ομάδες ε, της, ε, που έχουμε καταχωρήσει στον κατάλογο, όπως τα ΦΑΡΚ της Κολομβίας, το ΣΥΡΚ της ε, Σρι Λάνκα και το ΠΚΚ της Τουρκίας, που δεν ασκούν τρομοκρατικές ενέργειες στο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά χρησιμοποιούν τις χώρες της Ευρώπης για να συλλέγουν παράνομα χρήματα, για προπαγάνδα, για εκβιασμούς κτλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι τον Γκουαντάναμο. Θυμάστε ότι στα πλαίσια της εκθέσεώς μου του Νοεμβρίου του 2008 είχα προσκαλέσει το Συμβούλιο σε μια κινητοποίηση ταχυτάτη για να βοηθήσουμε τότε τον πρόεδρο, ο οποίος δεν είχε ακόμα ορκιστεί, να κλείσει το κέντρο του Γκουαντάναμο. Συζητήσαμε το θέμα και το Συμβούλιο πράγματι προσπάθησε να λειτουργήσει με ταχύτητα, με αποφασιστικότητα για να στηρίξει ουσιαστικά τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και να τον βοηθήσει όχι μόνο να κλείσει τον Γουαντάναμο, αλλά να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και έτσι ώστε αυτό το παράδειγμα το αμερικανικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να αλλάξει και να περάσει από μέτρα κάπως αυθαίρετα σε μέτρα τα οποία εδράζονται στο κράτος δικαίου όπως ακριβώς το κάναμε και πριν από τις τρομοκρατικές ενέργειες του Σεπτεμβρίου του 2011. Δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων υιοθέτησε μια κοινή ανακοίνωση μαζί με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Καταρχάς λέγεται ότι η ασφάλεια είναι σαφέστατα ευθύνη των κρατών μελών, αλλά είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε όλο και περισσότερο. Και ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παίρνει μέτρα τα οποία ε, να μην λαμβάνουν υπόψη το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες και πώς θα αντιδράσουν άλλες χώρες. Αυτό είναι συνέπεια της λογικής Σέγγεν, αν θέλετε. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε σχετικά με τον Γκουαντάναμο και όχι μόνο με τον Γκουαντάναμο η κυβέρνηση θα έλεγα έχει, των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αλλάξει εντελώς την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών φαινομένων. Και το Συμβούλιο προσπάθησε να συνεισφέρει στις εργασίες δύο task force, τα οποία δημιουργήθηκαν από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μία ασχολείται με τα θέματα των συνθήκων κράτησης και η δεύτερη με τα θέματα των μετακινήσεων και φύλαξης κατά τις μετακινήσεις των κρατουμένων. Προσπαθήσαμε εδώ να συνδέσουμε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το παραδοσιακό δίκαιο έτσι όπως λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ίδιος προσεκλήθη στην Washington στα μέσα Ιουλίου για να παρουσιάσω τις βασικές αρχές και να συνεργαστώ με τις δύο task force για την αλλαγή, πλήρη αλλαγή των μεθόδων που ακολουθούνται από τη ΣΥΠΑ. είναι σαφής η επιθυμία και των δύο πλευρών του Ατλαντικού να εμβαθύνουν τον διάλογό τους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Όταν πήγα στη Ουάσιγκτον, και είναι μια θα έλεγα εισαγωγή στη συζήτηση που θα κάνετε γύρω από την υπόθεση SWIFT, ε, είχε αλλάξει το κλίμα και ο, τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τους Αμερικανούς. Η σχέση μας είναι πολύ περισσότερο ουσιαστικά εταιρική είναι σχέση κατανόησης. Είναι μια ευκαιρία αυτή, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει σε επίπεδο συλλογής προσωπικών δεδομένων Ξέρετε ότι έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τι εργασίε τη ομάδα υψηλού επίπεδου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπω επίση και διαφόρων μέτρων που λαμβάνονται επιμέρου για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού φαινομένου. Τώρα για το SWIFT, δεν θα σα πω τώρα τίποτα, έτσι κι αλλιώ. θα κάνετε μια ειδική συζήτηση για το SWIFT και τότε ελπίζω να μου δώσετε την δυνατότητα να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Soy consciente έχω συνειδητοποιήσει, όπως όλοι μας, ότι το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι ένα ζήτημα μέγιστη ευαισθησίας και προτεραιότητας στις συζητήσεις στα κράτη-μέλη και στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις επίσης. Αλλά όπως υπενθύμισε ο συντονιστής για τα πολέμηση της τρομοκρατίας Ζήρ Κέρκοφ, έχουμε προγραμματίσει για τις 10.30 μία συνάντηση διμερούς χαρακτήρα των κοινοβουλευτικών επιτροπών ε, πολιτικών ελευθεριών και οικονομικών υποθέσεων και νομισματικών υποθέσεων υπό τη συμπροεδρία επιπλέον με την παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών ε, Sharon Bowles πράγμα που συνεπάγεται και σημαίνει ότι ζητώ κατανόηση από τα μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να θέσουν σε ιστερότερο χρονικό διάστημα τις ερωτήσεις ε, και τις παρατηρήσεις που σίγουρα προκαλεί η έκθεση, η εισήγηση του ε, αρμόδιου συντονιστή κατά πολέμησης τρομοκρατίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτείνω να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, το ακριβές αντίγραφο της εισήγησης που μόλις ακούσαμε τον κύριο Κέρκοφ με τέτοιο τρόπο ώστε θα μπορέσετε γραπτά να διατυπώσετε προς το γραφείο του συντονιστή καταπολέμησης της τρομοκρατίας τα σχόλια και τις ερωτήσεις που σας προκαλεί αυτή η εισήγησή του. Όμως επιπλέον σας προσκαλούμε ευμενώς να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο με την ε, Επιτροπή Κοινοβουλευτική, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στην επόμενη συνεδρίασή μας κατά τα τέλη του μήνα 29 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου και αν είναι στη διάθεσή μας ο συντονιστής θα είναι πρόσδεκτος, ώστε τότε, υστερότερα, να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί του μια συζήτηση που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον για όλα τα μέλη της κοινοβουλευτής μας Επιτροπής, διότι δυστυχώς αν τώρα ανοίγαμε γύρω παρεμβάσεων θα ήταν αδύνατο να έχουμε τη σημαντική συνεδρίαση μετά που θα ε, πρέπει να αρχίσει με τα μέλη της Επιτροπής ε, Νομισματικών και ε, Οικονομικών Υποθέσεων και κυρίως με τις αρχές που έχουν προσκληθεί για να μας εξηγήσουν το φάκελο την υπόθεση SWIFT που όπως ξέρετε εμπλέκει όχι μόνο τους ε, εκπροσώπους της ιδίας της υπηρεσίας SWIFT αλλά επίσης εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων κρατών μελών που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το χαρτοφυλάκιο. Προτείνω λοιπόν τώρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο να έχουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών για να προσέλθουν τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών και η πρόεδρος της αντίστοιχης Επιτροπής και να συνεχίσουμε αμέσως με το σημείο στην ημερήσια διάταξη για το, την υπόθεση SWIFT. Ευχαριστώ. Thank Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι να έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών, Επιτροπής ΕΚΟΝ και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπορώ να συμπροεδρεύσω αυτή τη συνεδρίαση με την πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ, κυρία Sharon Bowles. Τώρα, έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση ενώπιόν μας εδώ για να συζητήσουμε το θέμα της προσωρινής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ μετά από την ε, νέα ε, αρχιτεκτονική SWIFT. Και είχαμε σε αυτή την Επιτροπή τον ε, κύριο Μπαρό που παρουσίασε τις διάφορες τεχνικές ε, δυνατότητες ε, και εφαρμογές αυτής της αρχιτεκτονικής που συνεπάγεται και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την αρχιτεκτονική. Λόγω της ε, επίκαιρης κατάστασης των διαβουλεύσεων για την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ αυτό που θα κάνουμε είναι θα προχωρήσουμε σε δύο τμήματα στη συνεδρίασή μας. Το πρώτο τμήμα αυτής της συνεδρίασης θα είναι δημόσιου χαρακτήρα. Και θα έχουμε και ένα δεύτερο τμήμα που θα ακολουθήσει που θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτό σημαίνει, αυτά σημαίνουν ότι μόνο τα επίσημα μέλη ευρωβουλευτές και εντεταλμένοι αξιωματούχοι να συμμετάσχουν, θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν και να είναι παρόντες σε αυτό το δεύτερο τμήμα και κλεισμένων των θυρών της συνεδρίασής μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προσκαλέσει σε αυτή τη συνεδρίαση αρκετές αρχές και εκπροσώπους που θα παρέμβουν και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια ανοιχτή συζήτηση. Πρώτα λοιπόν θα έχουμε τον εκπρόσωπο του συστήματος SWIFT που θα παρέμβει για να μας ενημερώσει για τις αλλαγές και μεταβολές που υπάρχουν όσον αφορά την αρχιτεκτονική της δομής αυτής. Μετά θα έχουμε την αρχή, Βελγική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτικού Βίου σε σχέση με τα στοιχεία για το 2005 όσον αφορά τις αρχές των ΙΠΑ για την διαδικασία αυτή. Μετά θα έχουμε και πάλι τον υπεύθυνο συντονιστή καταπολέμησης της τρομοκρατίας κ. Ζίλντε Κέρκοφ και στο δεύτερο τμήμα και κλεισμένων των θυρών θα έχουμε μια συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αρμόδιους για τις διαπραγματεύσεις από πλευράς αυτών των δύο οργάνων. Υπενθυμίζω σε όλους σας ότι η νομική βάση που επελέγει από το Συμβούλιο <clears throat> στην πρόταση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι ο τρίτος πυλώνας. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν. Και σε σχέση με την υποχρέωση διαβούλευσης του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας και δεν έκανε χρήση το Συμβούλιο αυτής της δυνατότητας. Όμως εμείς από πλευράς Ευρωβουλής θα μπορούσαμε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς μας να αναλάβουμε πρωτοβουλία και να αποστείλουμε συστάσεις στους διαπραγματευτές πριν από την τελική σύναψη αυτής της ε, συμφωνίας. Και γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε ακριβώς και με βάση την έκθεσή μας ελπίζουμε ότι θα υπήρχε προετοιμασία σε σχέση με την διάσκεψη των Προέδρων του θέματος και έτσι καλωσορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών και την πρόεδρο, την πρόεδρο Sharon που δίνω τον λόγο άμεσα στην κυρία προτού προχωρήσουμε στον γύρο παρεμβάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία ήδη προαναφέρατε, διότι πρέπει να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, οι εισηγήσει και οι συζητήσεις. Θα ήθελα μόνο να πληροφορήσω τα μέλη ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρακολούθησα από την αρχή, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Το μέλημά μου ήταν να μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτές τις ε, αρχές που σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσες για την ε, Οικονομική Νομισματική Επιτροπή και Πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά τα θέματα έχουν ε, καλυφθεί, καλύπτονται πλέον. Προσβλέποντας το μέλλον τώρα, θα ήθελα να πω ότι ένα από τα θέματα που με απασχολούν τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε νομική βεβαιότητα και ασφάλεια σε σχέση με την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας. Και όχι μόνο νομική βεβαιότητα μεταξύ θεσμικών οργάνων και κυβερνήσεων, είναι αναγκαίο, πιστεύω πραγματικά, να υπάρχει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια για τον εμπορικό κόσμο, τους ε, ε, εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου που εμπλέκονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να είναι προηγούμενο για κάποια άλλα ζητήματα όσον αφορά τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις διεθνείς συναλλαγές και πληροφορίες. Αυτό θα ήθελα να πω αρχικά. Και παραδίδω τον λόγο για να παρέμβουν οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Thank ευχαριστώ κυρία Μπόλς. Και έτσι λοιπόν καλούμε να παρέμβει ο εκπρόσωπο SWIFT, ο κύριος Λάζαρο Κάμπος. Ήδη παρευρίσκεται. Παρακαλώ κύριε Κάμπος, μπορείτε να παρέμβετε. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Προφανώ, ένα αριθμό αριθμός ε, μελών έχουν προσκληθεί οι αρχές και θα θέλαμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος ε, Κάμπος, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους πρόεδρους κύριο Ροπεθαγγιλάρ και την κυρία Μπόρς για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση. Ο τίτλος της συζήτησης σήμερα επικεντρώνεται στις προτάσεις για μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα σαν αποτέλεσμα μιας νέας αρχιτεκτονικής SWIFT. Ωστόσο όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ευθύ εξ αρχής ότι η σημερινή συζήτηση δεν είναι για το SWIFT, είναι για το πώς η Ευρώπη προγραμματίζει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το SWIFT είναι ένα μόνο τμήμα και σκέλος που έχει επιπτώσεις αφορά από αυτή την ε, ε, προσπάθεια. Δεν θα έπρεπε με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζεται ε, από τους άλλους εμπλεκόμενους. Τα θέματα που συζητάμε έχουν οικουμενική σημασία και σπουδαιότητα. Αφορούν τους πολίτες, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και το παγκόσμιο σύστημα. Κατανοούμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα ήθελαν να συνεργαστούν ε, με τις οικονομικές αρχές των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συμμερίζονται στοιχεία που αποθηκεύονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ για το σύστημα SWIFT. Επίσης, μέσα στο πλαίσιο αυτό της ε, αρχιτεκτονικής SWIFT που είναι καταλήτης για αυτή τη νέα συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΕΠΑ, αυτή η νέα αρχιτεκτονική που μέχρι τα τέλη του έτους θα υλοποιηθεί, είχε το 2007 προαναγγελθεί ως με, με, μέρος των μέτρων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων για να υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες ε, των πελατών, διασφαλίζοντας και την ασφάλεια των δεδομένων. Τώρα σε σχέση με τα όσα έγιναν από την SWIFT και τα επιπλέον μέτρα τα οποία ελήφθησαν από τότε, υιοθετήθηκαν, εγκρίθηκαν από τις δημόσιες αρχές την ομάδα εργασίας 29 την Επιτροπή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου και τον υπατο εκπρόσωπο ανώτατο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατανοούμε την υποχρέωση να εξευρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και της κάλυψης των ε, αναγκών ασφάλειας ε, για τις ε, χώρες μας πάντα αναζητούσαμε να αναλυθούν όλες οι αναγκαίες ε, δράσεις για να μπορέσουν ε, οι στόχοι αυτοί να ευδοκιμήσουν. Έχει σημασία κλειδιού αυτό το SWIFT. Ε, βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος πληρωμών και συναλλαγών και εξοφλήσεων σε πολλές χώρες και σε διεθνές επίπεδο είναι ένα συμπλήρωμα του οικονομικού κόσμου, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικό αυτό όπως σήμερα, σε αυτές τις ταραχώδεις περιόδους που διανύουμε. Οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση των ε, επίκαιρων διαπραγματεύσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της δημοκρατίας, το έτοιμά μας θα ήταν να μην διακυβευτεί, να μην διακυβευθεί η προστασία που υφίσταται σήμερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, να μην διακυβευθεί η βεβαιότητα, η ασφάλεια όσον αφορά πλαίσιο και το ίσο δικαιο, ε, δικαιοδοτικά σύστημα, ισότιμο σύστημα το οποίο πρέπει να ισχύει για όλους όσους εμπλέκονται σε αυτές τις συναλλαγές. Όπως αναφέραμε είναι μια ε, ιδιωτική πρωτοβουλία που ε, συνεργάζονται σε αυτήν 9.000 τράπεζες, κεντρικές τράπεζες, οργανώσεις φορείς συμψηφισμού και εξοφλήσεων καθώς επίσης σε πάνω από 200 χώρες παγκόσμια. Το SWIFT επίσης έχει εποπτεία των, ε, των κεντρικών τραπεζών της ε, λέσχης των 10, διασφαλίζοντας ε, τον απόρριτο χαρακτήρα και διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην καρδιά των συναλλαγών μας. Γι' αυτό έχουμε ιδιαίτερε επιδόσεις στην προστασία αυτή. Και ταυτόχρονα έχουμε την διαβίβαση μέσω του δικτύου μας σε δύο κέντρα, σε δύο διαφορετικές υπήρους στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το πρώτο και το δεύτερο το κάνουμε αυτό για να αντιμετωπιστούν συστημικοί κίνδυνοι και να είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες και υπό τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις υπό το χειρότερο σενάριο. Θα υπάρξει και βελτίωση με ένα τρίτο ε, κέντρο στην ε, Ελβετία και θα υπάρχουν δύο ζώνες επεξεργασίας, μία στη ΣΥΠΑ, μία στην Ευρώπη. Αυτός ο, ε, θα έλεγα, διαχωρισμός σε δύο σκέλη θα επιτρέπει να διατηρούνται τα διευρωπαϊκά στοιχεία στην Ευρώπη Ευρώπη. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις, ε, τα μελήματα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε την ένταξη σε αυτές τις ε, ζώνες θυμόσαστε όπως αναφέρθηκε πιο πριν από τον Πρόεδρο ότι την τελευταία φορά που συμμετείχε σε μια κοινή συνεδρίαση η SWIFT ήταν τον Οκτώβριο 2006. Τότε η συζήτηση αφορούσε την υποχρεωτική ε, πρόσκληση από πλευρά των ΗΠΑ για την ε, μελλοντική λειτουργία στις ε, ΗΠΑ του κέντρου SWIFT. Σήμερα, χρόνια μετά, είμαστε εδώ παρόντες για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά υποστηρίζοντας το πρόγραμμα αυτό αναμένουμε οι ίδιες αρχές ε, σωστής ε, προστασίας ε, να ισχύουν και η ανάγκη να υπάρξει βεβαιότητα νομική, νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις. Οι ρήτρες ασφαλείας που θεσπίσαμε σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνουν τα εξής και τώρα υπογραμμίζονται ως βέλτιστες πρακτικές αυτές οι αρχές μέσα στο πλαίσιο αυτό. Έχουμε λοιπόν της ε, Σαπίνας που είναι περιορισμένες σε εύρος, προστατεύεται το πρόγραμμα αυτό, τα αιτήματα είναι στοχοθετημένα και βρίσκεται το πρόγραμμα αυτό σε συγκεκριμένες ε, ε, ε υπερπόντιες διαστάσεις. Και έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι για παράδειγμα μεγάλα χαρτοφυλάκια ε, τα οποία ε, μπορούν να, να εξαιρεθούν. Βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και διασφάλισης του απορρίτου οι αρχές των οικονομικών ε, των ΙΠΑ δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του SWIFT. Μόνο στοχοθετημένα αιτήματα μπορούν να διατυπώνονται και να ε, διαβιβάζονται, να διατίθενται τέτοια στοιχεία μόνο μέσα στο πλαίσιο ερευνών για την καταπολέμηση τρομοκρατίας η ε, πραγματική ε, ε, επιτήρηση και εποπτεία σε πραγματικό χρόνο που διασφαλίζεται, όπως επίσης και το πλαίσιο ασφαλείας είναι σημαντικά. Μέσα στα νέες ρυθμίσεις μεταξύ των αρχών των ΗΠΑ και Ευρώπης, οι ρήτες ασφαλείας δεν πρέπει να υποβιβάζονται ή να διακυβεύονται. Από την τελευταία φορά με την επιβεβαίωση της Επιτροπής από το Βέλγιο για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, και όσον αφορά και την αντίδρασή μας στις ε, σαπίνες των ΙΠΑ. Ε, ε, καλοχαιρετίζουμε αυτή την επιβεβαίωση της α, ε, συμμόρφωσης με τις αρχές αυτές της α, Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου, καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των όσων εμπλέκονται σε αυτά τα δίκτυα. Και να υπάρξουν ε, μηχανισμοί ευρωπαϊκοί για να επικουρούνται ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με θέματα συναφή με το SWIFT. Ολοκληρώνω και ε, ζητώ συγγνώμη για το ότι χρειάστηκα περισσότερα από πέντε λεπτά. Όπως ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου, αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη των δημόσιων αρχών να εξευρεθεί μια ορθή ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης της τρομοκρατίας αλλά ταυτόχρονα και της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει το SWIFT να συνεργάζεται με τον δημόσιο τομέα μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Από την άλλη πλευρά αναμένουμε ο δημόσιος τομέας να υποστηρίζει τον τομέα τον ε, ιδιωτικό και τις ανάγκες ε, της ε, διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο διαδρα... ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των όσων θα εμπλέκονται. Όλοι θα πρέπει να βρίσκονται υπό τις ίδιες αρχές και υπό την αντιμετώπιση από τις αρχές αυτές με τον ίδιο τρόπο ισότιμα θα πρέπει να μπορούμε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων σε εμά μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και των υποδομών που θα μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο από την δημιουργία του δικτύου μας του 1973 αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να ε, διακυβεύσει με κανένα τρόπο την αποτελεσματικότητα του SWIFT. Σήμερα για την, ε, το εύρος αυτό της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας οι έρευνες είναι στοχοθετημένες, ανεξάρτητα επιτηρούνται από ανεξάρτητες αρχές και έχουμε έτσι βελτιώσει την δυνατότητα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσα στην αρχιτεκτονική αυτή και την βελτίωση της στρατηγικής προσέγγισης. Διασφαλίζεται ότι στο τέλος θα πρέπει να παραμένουν αλόβητες ε, οι ε, διαδικασίες, οι διεργασίες αυτές. Θα πρέπει επίσης ε, από τις διεθνείς αρχές, με βάση διεθνείς αρχές να διέπονται αυτές οι συμφωνίες. Νέες προκλήσεις απαιτούν νέες λύσεις όμως και οι αρχές της ασφαλούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της νομικής ασφάλειας πρέπει να παραμένουν αλόβητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάμπος. Όπως είδατε, στην διαχείριση του ε, χρόνου θα παρακαλούμε ε, παρότι δεν είμαστε ακάμπτοι, ο κάθε συμμετέχον να τηρεί τον χρόνο που του δίνεται. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σε σχέση με τον χρόνο έγκαιρα μέχρι τις 12 ε, και 30 που έχουμε χρόνο τελικά. Τώρα ο κύριος Βίλεμ Ντε Μπόκελερ, πρόεδρος της Βελγικής Αρχής ε, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καλείστε να παρέμβετε, παρακαλώ. We were confronted Αντιμετωπίσαμε την υπόθεση SWIFT τον Ιούνιο του 2006, όταν η εφημερίδα New York Times απεκάλυψε ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην ε, διεκπαιρέωση προσωπικών δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα και που μπορούσε να αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες χωρίς καμία γνώση και χωρίς κανένα έλεγχο των ευρωπαϊκών ή βελγικών αρχών χωρίς κανένα έλεγχο τέλος των πολιτών. Τον Σεπτέμβριο του 2006 τότε η ε, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου εξέδωσε την πρώτη γνωμοδότηση σχετικά και τη στιγμή εκείνη είδαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη απόκληση, ένα μεγάλο πρόβλημα ανάμεσα στην Αμερικανική και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τουλάχιστον την νομοθεσία τη σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων που αφορά και το SWIFT. Και έτσι υπήρχε μια σύγκρουση δύο κόσμων νομοθετικού δυναμικού που δεν συμφωνούσε. Δεύτερη διαβούλευση, δεν υπήρχε καμία εμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή αλλά και η βελγική νομοθεσία για την, προσωπική, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εφαρμοστέα. Δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ αυτό. Αλλά ένα πρώτο νομικό πρόβλημα σημαντικό ήταν Ποιος φέρει την ευθύνη του ελέγχου για αυτές τις δράσεις και ποιος είναι υπεύθυνο για την παροχή των πληροφοριών αυτών από τις ευρωπαϊκές συναλλαγές, ε, των ευρωπαϊκών συναλλαγών δηλαδή, δηλαδή, στις αμερικανικές αρχές. Σε μια δεύτερη γνωμοδότηση, και αναφέρομαι στα έγγραφα τα οποία είναι στη διάθεσή σας και στην είσοδο της αίθουσας, στη δεύτερη γνωμοδότηση, τον Δεκέμβριο του 2006, απαντήσαμε σε ερώτηση της βελικής κυβερνήσεως, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματική προστασία των ε, Βέλγων πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, όσων δηλαδή αξιώνουν την προστασία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο μία λύση υπάρχει. Και δεν είναι βελγική λύση, είναι ευρωπαϊκή λύση. Και από τη στιγμή εκείνη, εμείς έχουμε ταχθεί υπέρ της αναζήτησης μιας λύσεως συνεργασίας που μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ε, συνθήκης ή και κάποια άλλη μορφή και που να συμφωνήσουν δηλαδή οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με τις ευρωπαϊκές αρχές. Και ε, είχαμε φτάσει την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που είχε γίνει με ανταλλαγή αλληλογραφίας, με διορισμό των αρμόδιων προσώπων. Είχε διεξαχθεί και μία έρευνα, νομίζω είχαν γίνει τα πρώτα σημαντικά βήματα. Ωστόσο δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Μια τρίτη γνωμοδότηση εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 2008, πέρσι, στις 9 Δεκεμβρίου, όπου εμείς εκεί ολοκληρώσαμε την διαδικασία για το SWIFT, όπου τονίζουμε και απαντώ και στην ερώτηση του Πρόεδρου της SWIFT, ότι δηλαδή επιβεβαιώσαμε ότι όντως η επιχείρηση SWIFT έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα των προσώπων. ώστε το κάθε πρόσωπο να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του και να χαίρει των ελευθεριών του. Το SWIFT δέχθηκε την ε, απόφαση της ε, Βελγικής Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και κάνει και τις σχετικές καταχωρήσεις στα σχετικά μητρώα. Η, τα δύο πιο σημαντικά συμπεράσματα και τα διδάγματα είναι δηλαδή πρώτο ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μόνες τους. Χρειάζεται να θεσπιστεί διεθνής μηχανισμός ελέγχου και είναι απαραίτητο ως ευρωπαϊκά νομοθετικά όργανα να εξασφαλίσουμε την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων μέσα στον κόσμο αυτό που ισχύει η αρχή της ελευθερίας της διακινήσεως των πληροφοριών. Και δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ε, ο πρώτος, το πρώτο καθήκον που έχουμε ως η Βελγική αλλά και η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι να προστατεύουμε και να εξασφαλίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό είναι και δίδαγμα αλλά κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσετε και εσείς για την εργασία που θα κάνετε, την νομοθετική εργασία δηλαδή, για την θέσπιση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών αρχών. Μην λησμονείτε λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που τηρήσατε το όριο χρόνου. Ε, θα ακολουθεί ο κύριος Πίτερ Χάσκινς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Πέντε λεπτά κύριε. Ζητήθηκε η γνώμη μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προβλεπόμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και τα SWIFT και δημοσίευσα κάποια σχόλια στις 3 Ιουλίου, οποία, τα οποία σχόλια είχαν σαν παραλήπτη την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα σχόλια αυτά ήταν όμως περιορισμένες κυκλοφορίες γιατί αναφερόντουσαν σε μια εντολή διαπραγμάτευσης, η οποία και αυτή από μόνη της είναι κατά κάποιο τρόπο εν μέρη απόρριτη απεστάλησαν μόνο τα όργανα τα οποία μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν δημοσιευθεί. Μπορώ όμως να σας δώσω μία περίληψη θα έλεγα των συζητήσεων μέχρι τώρα. Σαν δεύτερο σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική της SWIFT που ξεκίνησαν τις παρούσες διαπραγματεύσεις έχουν ενθαρρυνθεί και έχουν γίνει ευνοϊκώς δεκτό από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Έχουν σαν στόχο να θέσουν όλα τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών Αρχών. Έτσι, τα ευρωπαϊκά στάνταρτς για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιωτικά δεδομένα κτλ. θα πρέπει να εφαρμόζονται. Διαφορετικό είναι το θέμα από την υπόθεση PNR των προσωπικών στοιχείων, των επιβατών υπερατλαντικών πτήσεων. Η προτινόμενη συμφωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση SWIFT αφορά δεδομένα τα οποία δεν έχουν εδαφική θα έλεγα σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες καμία γιατί αναφέρονται σε ε, ενδοκινοτικές οικονομικές συναλλαγές και όχι σε οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα σχόλιά μου λοιπόν τον μήνα Ιούλιο εξέφρασα τις ανησυχίες μου σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα μιας τέτοιας συμφωνίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την παραβίαση της ιδιωτικότητας την οποία προκαλεί η πρόταση αυτή, όπως επίσης και την ύπαρξη ενός διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου στον συγκεκριμένο τομέα, ένα νομικό βλέσιο το οποίο ε, έχει σαν στόχο την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν εκφραστεί πάρα πολλές αμφιβολίες για τη νομική βάση της συμφωνίας. Γιατί αντίστοιχα κοινοτικά μέτρα τα οποία ισχύουν σήμερα βασίζονται στον λεγόμενο πρώτο πυλώνα. Όμως, σε αυτή τη φάση έχει σημασία να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις να λαμβάνουν υπόψη τους σοβαρά τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις ρήτρε ασφαλείας και να σέβονται φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα έτσι όπως ισχύουν και προστατεύονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ευρωπαϊκό έδαφος υπό ευρωπαϊκή δικαιοδοσία και οι εγγυήσει δεν θα πρέπει απλά να είναι περιορισμένες και το υπογραμμίζω αυτό, δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτά τα οποία θεωρούνται αποδεκτά όταν τα δεδομένα ελέγχονται από τις ελέγχονταν από τις Αμερικανικές αρχές. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε λοιπόν ποιος είναι ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και ποιος είναι ο μηχανισμός για το σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και των ατομικών στοιχείων. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα θαμελιώδη δικαιώματα δεν αφορούν μόνο την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα γιατί αυτή η κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων επηρεάζουν και άλλους τομείς των θεμελιωδών ελευθεριών και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να υπογραμμίσω ε, τα τέσσερα βασικά στοιχεία τα οποία ακολουθούν. Πρώτον, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την νομιμότητα και την αναλογικότητα των, των αμερικανικών απαιτήσεων στον συγκεκριμένο τομέα να δούμε υπάρχει σωστή στοχοθέτηση των ετοιμάτων πληροφόρησης των Αμερικανών. Αυτό θα πρέπει να ελέγχεται σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι αιτήσει αυτές για πληροφορίες να υφίστανται τον ίδιο έλεγχο, ακόμα και δικαστικό έλεγχο εάν χρειάζεται, όπως ακριβώς σημαίνει, συμβαίνει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα κρίσιμο το οποίο μέχρι τώρα θυμίζω στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων δεν έχει διευκρινιστεί. Ίσως ας πούμε να δούμε τι ισχύει στην περίπτωση της αμοιβαία νομικής βοήθειας στις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και στην περίπτωση όπου υπάρχουν παραβιάσεις να υπάρχει η δυνατότητα αποζημιώσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα επίσης δικαστικής αποκατάστασης πέραν της διοικητικής. Αυτό δεν είναι μόνο μια απέτηση σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά είναι μια γενικότερη απέτηση η οποία προέρχεται από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβεβαιώνεται από την ευρωπαϊκή νομολογία σε περιπτώσεις ε, όπως η γνωστή υπόθεση Κάρντι σχετικά με κάποιους Ταλιμπάν νομίζω ε, δείχνει ότι οι μηχανισμοί αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνονται όχι μόνο στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας αλλά και να καλύπτουν και την ίδια SWIFT, η οποία SWIFT θα πρέπει να είναι σε θέση να αμφισβητήσει σε δικαστικό ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβολικές απαιτήσει των Αμερικανών. Τρίτον, περαιτέρω ε, θα έλεγα κατανομή των στοιχείων αυτών και με άλλες υπηρεσίες και με άλλες χώρες θα πρέπει να ε, υπόκειται ακριβώς στις ρυθμίσεις που έχει προτείνει το Συμβούλιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τις ενδοκινοτικές συναλλαγές. Θα ήταν παράδοξο να δεχθεί για τις εξωτερικές υπηρεσίες ξένων χωρών ένα καθεστώς λιγότερο αυστηρό από ό,τι δεχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ίδια, για τα, ίδια τα όργανα τα κοινοτικά. Θα πρέπει επίσης το SWIFT, τα πιστοτικά ιδρύματα και οι μηχανισμοί ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο από τη διεθνή αυτή συμφωνία. Ο ανεξάρτητος έλεγχος είναι βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξέταση των αναφορών και παραπώνων, και ακριβώς αυτό το πλαίσιο να μου επιτρέψετε να τονίσω ότι οι περιοδικές ρυθμίσεις και έλεγχοι της κατάστασης ήταν τμήμα των υπαρχουσών συμφωνιών, είναι τμήμα των οδηγιών που ισχύουν σήμερα και θα πρέπει να είναι τμήμα των συμπερασμάτων στα οποία θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες εξηγήσεις. Ευχαριστώ κύριε Χάστινγκς. Περνάμε τώρα στα υποδιαπραγμάτευση θα έλεγα ευρωπαϊκά όργανα. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φάουλ. Σας ευχαριστώ. Θα εξηγήσω τι έχει ήδη συμβεί, τι γίνεται και τι ελπίζουμε να συμβεί στο μέλλον. Σήμερα η κατάσταση έχει ως εξής. Μετά από, την, από τις αποκαλύψεις για το τι έκανε η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, τι έκαναν και άλλοι φορείς, ξαφνικά ξεπίδησε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, διοχετεύονταν δεδομένα για Ευρωπαίους πολίτες στις Αμερικανικές αρχές και εκτός της, ε, των εταιριών που αναμειγνύονταν και των Αμερικανικών αρχών, ουδής εγνώριζε τίποτε. Ε, η κοινή γνώμη ανησύχησε βέβαια και δικαίως. Και τέθηκε το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο υψηλότερο επίπεδο, και ιδίω από έναν Πρωθυπουργό ο οποίο είναι σήμερα Ευρωβουλευτή, ζητήθηκε λοιπόν από το υψηλότερο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει και να βρει τρόπο να ε, κάνει συμβατά τα προβλεπόμενα από τη δική μας νομοθεσία με αυτά που ζητεί μια άλλη ξένη χώρα χωρίς να ε, βρεθούν τελικά τα προσωπικά δεδομένα εν κενό κάπου υπεράνω του Ατλαντικού. Το κάναμε αυτό με πλήρη ενημέρωση και των κοινοβουλευτικών σας επιτροπών. Διαπραγματευθήκαμε έναν αριθμό ρυθμίσεων με την ε, Αμερικανική κυβέρνηση που κατά τη γνώμη μας είναι ικανοποιητικέ που αναλύθηκαν βεβαίως και από τον ε, ε δικαστή κύριο Μπεκελάρ, ο οποίος θα μας πει μετά νομίζω ε, που κατέληξε και μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη βάση χωρίς όμως η βάση αυτή να είναι ικανοποιητική, διότι δεν είναι επίσημη δεσμευτική συμφωνία. Και έγινε βέβαια υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές υπό τις οποίες θέλουμε τώρα, λόγω της απόφασης της SWIFT να μεταθέσει ορισμένα από τα δεδομένα από τις, ΗΠΑ από, την... Ε, από τις Ηνωμένες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι βρισκόμαστε σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, διότι ναι μεν σήμερα οι πιο πιστικές αναλύσεις μας λένε ότι είναι θέμα του τρίτου πυλώνα, ελπίζουμε όμως, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η συνθήκη της Αβώνας θα τεθεί σε ισχύ, ότι ε, θα πάψουν να ισχύουν οι πυλώνες και ότι θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο καθεστώς το οποίο θα επιτρέπει βεβαίως και πολύ πληρέστερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν ένα προσωρινό πρόβλημα, το οποίο είναι πώς θα περάσουμε από τη σημερινή κατάσταση στην αυριανή, προβλέποντας μια διεθνή συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην SWIFT να συνεχίσει τις απόλυτα νόμιμες άλλωστε και θεμητές δραστηριότητές της και οι τράπεζες που είναι γνωστόν ότι έχουν βέβαια και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν την περίοδο αυτή, να μπορέσουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες των. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα λόγω και της απόφασης της SWIFT να μεταθέσει τις βάσεις δεδομένων της. Α, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι βέβαια για την ενέργεια αυτή. Αυτό που προτείναμε και που το υποστήριξε ομόφωνα το Συμβούλιο Υπουργών είναι ένας αριθμός διαπραγματευτικών κριτηρίων σχετικά με μια πολύ βραχυπρόθεσμη προσωρινή συμφωνία η οποία θα προσφέρει επαρκής, επαρκή προστασία και τους απαραίτητους μηχανισμούς εποπτείας. Και αυτό για την διάρκεια ανάμεσα στην θέση σε ισχύ της συμφωνίας αυτής και στην υπογραφή νέα συμφωνία που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει πολύ γρήγορα όταν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Εγώ πάντως μπορώ να λάβω τη δέσμευση και εκ μέρου τη Κομισιόν και του Επιτρόπου Ζακ Μπαρό ότι όταν η συνθήκη τη Λισαβόνα θα τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει νέες, νέα πρόταση διαπραγματευτικής εντολή στο Συμβούλιο για να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση συμφωνίας που θα συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα από την συνθήκη της Λισαβόνας και με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Κάτι που πρέπει να ε, θυμόμαστε είναι ότι πρόκειται για αντιτρομοκρατική δραστηριότητα. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια των ΗΠΑ, είναι και η δική μας ασφάλεια που διακυβεύεται. Η ασφάλεια των χωρών μελών μας, του εδάφους μας, των πολιτών μας. Οι πληροφορίες που δίνονται με πολύ συγκεκριμένους και περιορισμένους όρους, όπως εξήγησε ο κ. στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, γίνεται με βάση μια ανάλυση που κάνουν οι αρμόδιες αρχές των χωρών μελών μας, οι οποίες δέχθηκαν την ανάλυση αυτή και τη θεωρούν χρήσιμη και τι προφορίες δηλαδή αυτέ, χρήσιμε για την καταπολέμηση τη δημοκρατίας και εδώ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που κάνουμε μοναχά για χάρη των ΗΠΑ, είναι κάτι το οποίο γίνεται και προ το δικό μα συμφέρον. Και είναι βέβαια σημαντικό, όπω είπε και ο κύριος Κάμπος στη SWIFT, ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε οι επιχειρήσει να βρεθούν σε κενό, να βρεθούν μετέωρε σε ένα χώρο εκτός δικής μας νομοθετικής αρμοδιότητας και εκτός νομοθετικής αρμοδιότητας των ΗΠΑ. Πρέπει αντίθετα να βρούμε λύσει που θα επιτρέψουν στα γρανάζια και στου τροχούς του εμπορίου να συνεχίσουν να κυλούν και να κινούνται. Να επιτρέψουμε δηλαδή την απαραίτητη ροή των πληροφοριών που θα επιτρέψει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φόλ. Για τον πρώτο αυτό γύρο λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στον ε, ε, εκπρόσωπο της Προεδρίας, κύριο Χένιγκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σας. Εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε τα περισσότερα από αυτά τα οποία θα ήθελα να πω και θα είμαι συντομότερο των πέντε λεπτών και έτσι θα κερδίσετε κάποιο χρόνο. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αυτά τα οποία σαν Προεδρία έχουμε κάνει μέχρι τώρα και χωρίς να έχουμε φυσικά γνώση των θεμάτων όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι τον Ιούνιο φέτος ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και όπως γνωρίζετε η Σουηδία και η Σουηδική Προεδρία έχουν σαφείς ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των στοιχείων αυτών, κάτι το οποίο συνιστά σουηδική παράδοση θα έλεγα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε περισσότερα από τα σημεία, τα περισσότερα από τα σημεία περιλαμβάνει η έκθεση την οποία παρουσίασε ο κ. Χούστινγκς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Κάνουμε δεκτά τα περισσότερα από τα σημεία αυτά λοιπόν. Αν και συνεχίζουμε τυπικά τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι μετά από την υιοθέτηση της εντολής αυτής στο Συμβούλιο στα τέλη του μηνός Ιουλίου, είχαμε δύο διαπραγματευτικές συνόδους με τους Αμερικανούς από κοινού. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αυτές και τον μήνα Σεπτέμβριο με στόχο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν στα πλαίσια τουλάχιστον των χρονικών προσθεσμιών που αφορούν τη Σουηδική Προεδρία. Η Σουηδία και η Σουηδική Προεδρία, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζουν ότι πριν από την αλλαγή της νομικής βάσης θα έχει μεσολαβήσει η υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας, το ελπίζουμε αυτό, και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις στα πλαίσια μιας νέας μονιμότερης συμφωνίας η οποία θα εμπλέκει πλήρως θεσμικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γέφυρα χρονικά, η οποία να έχει μέγιστη διάρκεια ισχύω ένα δωδεκάμινο, δηλαδή συντομότερη χρονική διάρκεια και να μπορέσουμε αν είναι δυνατόν στην καλύτερη περίπτωση να την αντικαταστήσουμε τη συμφωνία αυτή και πριν από το τέλος του 12 μήνου. Η Σουηδική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέλλον του καθεστώτος αυτού μετά την υιοθέτηση της συνθήκης. Πότε μπορεί να ξεκινήσει μια νέα διαπραγματευτική εντολή και σύμφωνα με τον κύριο Μπαρό θα ξεκινήσει αμέσως μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας όταν γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει τώρα για λεπτομέρειες περισσότερες και για το ποιος αναλαμβάνει την διαπραγμάτευση Αυτά θα τα συζητήσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ κύριε Χένιγκεν. Έχουν ζητήσει εννέα μέλη της Επιτροπής τον λόγο. Και ο, ο κύριος Ζίλντο Κερκόβε έχει ζητήσει και αυτό το λόγο. Ο εκπρόσωπος της ε, Συντονιστικής Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά από τον κύριο Ντοκερκόβ. Θα ήθελα ακριβώς να ξεκινήσω σαν συντονιστής της καταπολέμησης ε, της τρομοκρατίας και να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φάουλ. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των μεθόδων χρηματοδότησης, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και παρακολουθείται από πολύ κοντά όχι μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μας εποφελούνται του συστήματος αυτού. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη το σύστημα αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεύτερον, η έκθεση De Brugger απέδειξε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποδέχονται και εφαρμόζουν πλήρως τις ανηλυμένες τους υποχρεώσεις. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί γίνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολες. Τρίτον, η αλλαγή αρχιτεκτονικής του SWIFT οδηγεί σε μια επανεξισορρόπηση των σχέσεων. Όπως είπε ο Φόουλ, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες διαπραγματεύσεις, τα δεδομένα βρίσκονται στις Ηνωμένε Πολιτείες, τώρα βρίσκονται στην Ευρώπη και ακριβώς διαπραγματευόμεθα σε επίπεδο εταιρικό πλέον. Και αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πρόσβαση πιο αποτελεσματική στο ίδιο το σύστημα. Τέταρτο στοιχείο, μια νομική συμφωνία η οποία να βασίζεται στο άρθρο 24 της συνθήκης θα καλύψει νομικά και μάλιστα με δεσμευτικό τρόπο τις εγγυήσει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν παρά σε μονομερές επίπεδο αντικείμενο προστασίας από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Γι' αυτό λοιπόν η διαπραγματευτική εντολή της Προεδρίας και της Επιτροπής είναι ισόρροπη και απαιτητική προϋποθέτει αυστηρά συστήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θυμίζω ότι γίνεται μια παράλληλη συζήτηση για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων ανάμεσα στις ΗΠΑ και, στις Ηνωμένες... και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία και εδώ. Δεύτερο στοιχείο, και έχει σημασία αυτό αφού άκουσα αυτά που είπε ο κ. Χάστινγκς, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στο πλαίσιο το ακριβές μέσα στο οποίο λειτουργεί η συμφωνία αυτή και εδώ το πλαίσιο αυτό θα μπορεί να είναι και καλυπτόμενο από δικαστικές αποφάσεις. Τρίτον, η διάρκεια της συμφωνίας και η ισχύ της συμφωνίας μέσα στο χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Είναι τέτοια που επιτρέπει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε στο μέλλον είτε να συνεχιστεί η ισχύ του παρόντος συστήματος, είτε να υπάρξει ένα νέο σύστημα σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι έχουμε και μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών σε λίγη ώρα και θα παραμείνει χώρος για συζήτηση και στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής και κλεισμένων των θυρών. Έχουν ζητήσει ακόμα 12 μέλη το λόγο. Θα πρέπει να κλείσουμε τη λίστα πλέον και θα ήθελα να σας προτείνω για να έχουμε κάποιο λογικό χρόνο να συνεχίσουμε να περιοριστεί κάθε μέλος σε μια δίλεπτη παρουσίαση ερώτηση. Δίλεπτη. 1,5 λεπτό, όχι καν, ούτε καν δύο λεπτά. 1,5 λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Λαμπρινίδης έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους. Σε 1,5 λεπτό, την από τέσσερα σημεία. Ο Φάουλ παρεδέχθη κάτι το πολύ σημαντικό. Τι μας είπε ο Φάουλ. Ότι στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει σαν υπεργολάβο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή, στέλνουμε τα στοιχεία στις Ηνωμένε Πολιτείε, αναλύουν τα στοιχεία και μετά μας ε, αναφέρουν πού είναι τα προβλήματα, αν υπάρχουν προβλήματα. Και φυσικά η νομική βάση είναι αυτή η οποία είναι. Δεύτερο, ο εκπρόσωπος του SWIFT ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για τις αιτήσει των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα τρομοκρατίας μόνο και μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλοι είπαν εδώ ότι πάρα πολύ ωραία έχουμε μια καλύτερη ισορροπία γιατί διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μια ιδιωτική εταιρεία. Το ερώτημά μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξής. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτών, αυτοί οι άξονες και οι ρήτρε προστασίας διατηρούνται όπως ακριβώς γινόταν αυτό στο παρελθόν. Και αν ναι, τότε γιατί ξαφνικά ε, γιορτάζουμε θα έλεγα τις περισσότερες αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε αποκτήσει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη ερώτηση. Προς τη Σουηδική Προεδρία. Σέβομαι την Προεδρία αυτή, αλλά έχω επίσης και σεβασμό απέραντο προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπατε ότι και εσείς στη χώρα σας σέβεστε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ιδιωτικά δεδομένα. Να πω όμως ότι πολλές συζητήσεις που γίνονται για τον έλεγχο στο διαδίκτυο και νόμοι οι οποίοι ισχύουν σε διάφορες χώρες ε, είναι νόμοι οι οποίοι βασίζονται στη σουηδική εμπειρία. Το ερώτημά μου είναι το εξής λοιπόν. Θέλετε να βάλετε τον ίδιο βαθμό ελέγχου και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή θα θέλετε να εφαρμόσετε τα επίπεδα ελέγχου τα οποία εφαρμόζεται στον έλεγχο του διαδικτύου. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το 1,5 λεπτό, αλλά πάντως δικαίωμα των βουλευτών να θέτουν ερωτήσεις και όχι να κάθονται απλώ εδώ και να ακούν ομιλίες. Λοιπόν, πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί. Γιατί Πρώτα ορίζουν οι κυβερνήσεις τι επιθυμούν να κάνουν και μετά ρωτάνε τον κόσμο αν μπορούν να πάρουν τις προφορίες αυτές. Ενώ σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να, είναι, να βασίζεται η προσπάθεια αυτή στην συμπτωματική διαθεσιμότητα ορισμένων πληροφοριών. Και γι' αυτό συμφωνώ και με τον Σταύρο στις ερωτήσεις που έκανε. Δεύτερο, φαίνεται να υπάρχουν ε, απόψει σχετικά με την νομική βάση. Φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και στη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Και θα συστήσω στην παρούσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ζητήσουμε μια ανάλυση από ε, μια εξωτερική υπηρεσία, από ένα εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Για την περίπτωση P&R ζήτησε το Κοινοβούλιο τέτοια ανάλυση εξωτερική. Επίσης θεωρώ ότι όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ε, δημόσιο κτήμα. Και γι' αυτό ρωτώ, γιατί γίνεται και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση και όχι να βρίσκονται τα έγγραφα μονάχα φυλασσόμενα σε ε, ειδική αίθουσα και μόνο πρόσιτα σε ορισμένους βουλευτές. Θα ρωτήσω λοιπόν, αν φού δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, γιατί δεν το καθιστάτε δημόσιο. Όλο, τα όλα τα εγγραφά δηλαδή. Και τέλο ένα πράγμα που δεν κατανοώ είναι, λίγου μήνε πριν υποτίθεται, λίγου μήνε μετά μάλλον, υποτίθεται ελπίζουμε ότι θα, μπει σε, θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα και θα έχουμε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο. Εάν πραγματικά οι Ευρωπαϊκέ κυβερνήσει δεσμεύονται υπέρ τη δημοκρατία, γιατί αυτή η εντολή δεν έγινε δημόσια και να έχει τεθεί υπό την έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το λιγότερο. Ο κύριος Λουί Μισελ. Είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί η συνάδελφο πράγματι έθεσε τι περισσότερε από τι ερωτήσει που θα ήθελα και εγώ ίδιο να θέσω. Υπάρχουν πάρα πολλά αγκάθια τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια τη συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να χειροτερεύσουμε την εικόνα μια εταιρεία η οποία φαίνεται ότι εργάστηκε μέχρι τώρα σεβόμενη τα καλύτερα δυνατά επίπεδα δεν θα πρέπει να καταστρέψει